Έχει το λόγο η κυρία ε, Σενιάλοβα. Το λόγο. Και εάν θέλετε να αποχωρήσετε αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να το πράξετε ταχαίως και σιωπηλός. Κυρία Σενιάλοβα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει ενώ ορισμένη αποχωρείται από την αίθουσα. Μια συζήτηση η οποία έρχεται μετά από την έγκριση στις 2 Μαρτίου εξ ονόματος του Συμβουλίου τις θέσεις του σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τον κανονισμό για τις απαιτήσει έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί τμήμα πρωτοβουλειών, απότερο στόχος των οποίων είναι να χρησιμοποιηθεί το σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην υπηρεσία 112 στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια υπηρεσία την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν όλοι οι καταναλωτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη είχαν αποφασίσει ότι θα πρέπει το σύστημα e-call να χρησιμοποιείται σε όλα τα οχήματα υποχρεωτικά και μάλιστα από τον Οκτώβριο του 2017. Θα προβλέπετε λοιπόν μια πανευρωπαϊκή υποδομή προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κείμενο αυτό συμπληρώνει το αρχικό κείμενο και αναφέρεται συγκεκριμένα στι απαιτήσει έγκριση τύπου, προκειμένου να μπορεί να ενσωματώνεται το σύστημα σε όλα τα νέα οχήματα. Αναφερόμαστε κυρίω εδώ πέρα σε επιβατηγά οχήματα και σε ελαφρά φορτηγά και από την 1η Μαρτίου του 2018 θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τον μηχανισμό e-call προκειμένου σε περίπτωση ατυχήματο να μπορεί αυτόματα χειρονακτικά να ενεργοποιείται ο αριθμό 112. Στο παρελθόν, είχαμε επιμείνει ότι ε, υπήρξε μια σημαντική καθυστέρηση όσον αφορά την εθελούσια εφαρμογή του συστήματος αυτού. Πλέον όμως ε, στην πρόταση κανονισμού και έπειτα και στην απόφαση του 2012 είχαμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση προκειμένου η υπηρεσία 112 να καταστεί δημόσια υποχρεωτική υπηρεσία. Τον Ιούνιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα κείμενο βάσει το οποίο εργαστήκαμε και η Επιτροπή Προστασία του Καταναλωτών και Εσωτερική Αγορά, Επιτροπή Μεταφορών, Επιτροπή Βιομηχανία, Επιτροπή Ενέργεια και Βιομηχανία, η Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων υποστήριξαν ότι θα πρέπει το σύστημα αυτό να υποχρεωτικό και να ενσωματώνεται υποχρεωτικά σε όλα τα νέα οχήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει ισχυτέ, του συντάκτε γνωμοδότηση και όλου όσοι συμμετείχανε σε αυτή την όλη εργασία που κάναμε προκειμένου να καταφέρουμε να διευκρινίσουμε, να αποσαφηνίσουμε περισσότερο το κείμενο. Το Φεβρουάριο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και κατά αυτόν τον τρόπο δόθηκε και μία εντολή διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίησαν πολλές φορές το κείμενο και Κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2014 έλαβαν χώρα τρει τριμερεί διάλογοι, καθώ επίση και πολλέ συζητήσει ε, εργασία, προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε τελικά σε μια διοργανική συμφωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο τη Ιταλική Προεδρία αλλά και τον εκπρόσωπο τη Λετωνική Προεδρία για την πολύ επικοδομητική του συνεργασία. Καταφέραμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταλήξουμε συμβαστική λύση που έχετε ενώπιον σα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να καταθέσει συγκεκριμένε τροπολογίε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Για παράδειγμα, είπαμε ότι θα πρέπει να γίνεται μια συγκεκριμένη αναφορά στον αριθμό κλίση έκτατη ανάγκη 112, ότι θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με τα συστήματα ραδιοπλοήγησης. Είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον μία έκθεση προκειμένου να γίνει μία καλύτερη αξιολόγηση των νέων υπηρεσιών προστιθέμενων υπηρεσιών επιπλέον αξίες, προστιθέμενες αξίες, προκειμένου να καταφέρουμε να καταστήσουμε το σύστημα αυτό ακόμα πιο αποδοτικό και να μπορέσει να συνεργαστεί δικό τομέα. Στα πλαίσια του νέου αυτού κειμένου προστατεύουμε σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή. Αυτό το στοιχείο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτέλεσε σημαντικό μας μέλημα από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Καταφέραμε λοιπόν να δημιουργήσουμε σαφείς κανόνες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών αυτών δεδομένων. Τα οχήματα τα οποία θα έχουν έναν σωματωμένο σύστημα e-call δεν θα αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ανείχνευσης και παρακολούθησης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι ανενεργό και να χρησιμοποιείται μόνο όταν ενεργοποιείται το σύστημα κλήση. Όλα τα δεδομένα τα οποία θα μεταφέρονται από το όχημα προ τα κέντρα επεξεργασία τη κλήση έκτακτη ανάγκη θα μεταφέρουν τα ελάχιστα μόνο δεδομένα τα οποία απαιτούνται για να εντοπιστεί το όχημα και ο χώρο του ατυχήματο. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται η εσωτερική μνήμη του συστήματος να καταγράφει όλα αυτά τα δεδομένα. Επίσης, η ημερομηνία θέση σε ισχύ του κανονισμού έχει μετατεθεί. Προβλέπεται ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με πάρα πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και γι' αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη ζήτησαν περισσότερο χρόνο προκειμένου να δημιουργήσουν μαζί με αυτούς τους τρίτους φορείς απαραίτητες υποδομές. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σα ζητώ να εγκρίνετε το κείμενο αυτό χωρί περαιτέρω τροποποίηση. Έχουμε μπροστά μα μια συμφωνία διοργανική που αποτελεί προτεραιότητα τη Επιτροπή ε, Εσωτερική Αγορά και αποτελούσε ουσιαστικά την έκβαση τη πρώτη αυτή εντολή που μου είχε δοθεί σε επίπεδο πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η συμβαστική λύση που έχουμε μπροστά σα πραγματικά αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται στι προσδοκίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια. Τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, Φιλ Χόγκαν, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Συχνάλοβα της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς για τις ακούραστες προσπάθειές της. Ε, Επιτρόπος ε, ε, που έχει το θέμα αυτό στην υπευθυνότητα, στην ευθύνη της δεν είναι εδώ, οπότε αναλαμβάνω εγώ το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις επιτροπές που αναμίχθηκαν ε, όχι μόνο την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, διότι συνσέφεραν πάρα πολύ θετικά. Η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Ε, ήδη έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να συμβαίνουν οδικά ατυχήματα και αρκετά συχνά. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ε, θα ειδοποιηθούν οι κατάλληλες αρχές το συντομότερο δυνατό και με τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Αυτό ε, κάνει μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά τα θύματα. Το e-call είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο αυτόματα ενημερώνει τις, ε, ε, τους αρμόδιους φορείς για το ατύχημα και δίνει αρκετές λεπτομέρειες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε δραστικά το χρόνο παρέμβασης, επέμβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε αυτή την ιδέα πριν από ένα χρόνο, τον Απρίλιο του 2014, το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την απόφαση να τεθεί σε ισχύ το σύστημα e και σήμερα μπορείτε πλέον να εγκρίνετε τον κανονισμό που θα επιτρέψει τη λειτουργία του συστήματος. Πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα ισορροπημένο κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε ζωτικό ρόλο για την στήριξη αυτής της προσπάθειας το κείμενο δεν αγνοεί το γεγονό ότι υπάρχουν ήδη στην αγορά ιδιωτικά συστήματα που, των οποίων επιτελεσματικότητα έχει αποδεχθεί. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμή του κανονισμού θα καταστήσει υποχρεωτική την ε, εγκατάσταση αυτού του συστήματος σε όλα τα οχήματα στο μέλλον. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται υπόψη και οι ανησυχίε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και του απορρίτου. Γι' αυτό το λόγο, ε, οι πληροφορίε που μεταδίδονται είναι μόνο οι απολύτω απαραίτητε και οι πληροφορίες αυτές φεύγουν από το αυτοκίνητο μόνο όταν συμβαίνει ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα και ε, δεν παραμένουν αποθηκευμένες στο όχημα. Με αυτόν τον τρόπο τα, οι, οι κλείς αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθηθεί κάποιος. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την, ε, προ, τη συνεισφορά της ε, Επιτροπής Ατομικών Ελευθεριών. Τώρα, κατανοώ βέβαια και την ε, ε ανυπομονησία σας ε, να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό ήδη από το 2018. Ε, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχουν οι πολιτικές ομάδες και πρώτος ο κύριος Κάρλος Κουέλιο, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παρακαλώ, για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σενάλοβα για την έκθεσή της. Μετά από τρεις τρίλογους και συνεδριάσεις εργασίας μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο έκθεσης για αυτό το θέμα το οποίο έχει ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2003. Το κείμενο αυτό το οποίο θα ψηφιστεί λοιπόν αύριο στην Ολομέλεια αντικατοπτρίζει μια πραγματική προσθέμενη αξία για την ασφάλεια στους οδικούς άξονες και για τη ζωή των πολιτών μας. Το σύστημα e-call σώζει ζωές. Σώζει αυτούς που χάνουν τη ζωή τους και γλιτών και τις οικογένειες από την απώλεια των ε, οικείων τους με ένα νούμερο, το 112, το οποίο μπορεί να κληθεί αυτόματα από το όχημα. Σε περίπτωση που είναι που λαμβάνει η χώρα ένα σοβαρό ατύχημα υπάρχει η αυτόματη κλίση προς μια υπηρεσία που διαβιβάζει τα απαραίτητα στοιχεία για το όχημα και τους επιβάτες και επιτρέπει την ταχύτερη έλευση των σωστικών συνεργείων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος. Είναι λοιπόν <clears throat> απαραίτητο αυτή η νομοθεσία σε σχέση με το e-call για να εγκατασταθεί αυτό το σύστημα αυτόματης κλίσης στο 112 είναι ένα πολύ καλό σύστημα, καλή απόδειξη του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε συστήματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά όσο η μείωση των θανάτων στους δρόμους και η καλύτερη αρρωγή στα θύματα των οδικών ατυχημάτων. Είναι δωρεάν υπηρεσία του ECOL, είναι ασφαλής, μπορεί να λειτουργεί σε όλα τα κάτι και σέβεται αυστηρά τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος e-call από το Μάρτιο του 2018 θα είναι υποχρεωτική και με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί σημαντικά η ασφάλεια στους δρόμους και η προστασία των πολιτών. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει κυρία Γκέπχαρ για ένα λεπτό, για ένα μισή λεπτό, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε... Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αυτούς που ενεπλάξαν στην τόσο οικοδομητική εργασία για το σύστημα e-call το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει όλους. Και εμείς φυσικά ως σοσιαλδημοκράτες θα υποστηρίξουμε αυτό το κείμενο συμβασμού. Για μας σοσιαλδημοκράτες ήταν απαραίτητα απαραίτητον να εξασφαλίσουμε ότι η βοήθεια ε, θα έρθει μετά από ένα τύχημα το ταχύτερο δυνατό. Γι' αυτό το σύστημα e-call είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ένα πρόβλημα είχε διαγραφεί από την αρχή με το σύστημα αυτό η υποστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό ήταν από τα κέρια ερωτήματα τα οποία τέθηκαν σε συζήτηση και ήταν ένα θέμα αμφιλεγόμενο στον τομέα αυτό. Πιστεύω όμως ότι η λύση η οποία, η οποία επετεύχθη για το λεγόμενο υπνώτον σύστημα είναι η καλύτερη λύση. Με το σύστημα αυτό δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να παρακολουθηθεί η διαδρομή ενός οχήματος. Υπάρχουν ήδη πολλά ιδιωτικά συστήματα τα οποία λειτουργούν και τα οποία ήδη ε, έχουν σαν στόχο να δίδουν στοιχεία για την ε, ιατρική κατάσταση του οδηγού και τα λοιπά. Όχι, δεν θέλουμε εμείς ένα τέτοιο σύστημα, θέλουμε απλώς ένα σύστημα το οποίο ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό της ε, δυνάμεις διάσωσης και επομένως δίνει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που έχει λάβει η χώρα ένα ατύχημα, σε ποια περιοχή και αυτό εξασφαλίζει ότι η αρρωγή θα έρθει το ταχύτερο δυνατόν. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό έχουμε επιτύχει κάτι πολύ θετικό, εξασφαλίζουμε την προστασία δεδομένων αλλά και την ταχύτατη παροχή βοήθειας που είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Πανμποσού έχει τώρα το λόγο εξ ονόματος του ECR για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Δεκέμβριο, στα πλαίσια της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ, καταλήξαμε σε μια συμφωνία όσον αφορά το σύστημα e-call και μετά από τέσσερις μήνες, ως σκιώδη ηγήτρια του ECR, Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το νέο αυτοκείμενο που έχουμε ενώπιόν μας και θεωρώ πλέον ότι μπορούμε να επισημοποιήσουμε αυτό το νέο κανονισμό. Όλο και περισσότερο χάνουμε συμπολίτε μα εξαιτία των τροχαίων ατυχημάτων και χάρη στο νέο αυτό σύστημα e-call θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει στο παρελθόν πάρα πολλέ ανθρώπινε ζωέ. Το σύστημα αυτό θα σώσει όμω στο μέλλον πολλέ ανθρώπινε ζωέ. Όπω ακούσατε, υπάρχει μια αυτόματη διασύνδεση με τα κέντρα λήψη κλήσεων έκτακτη ανάγκη και νομίζω ότι αυτά τα λίγα λεπτά θα μα βοηθήσουν πραγματικά να σώσουμε όλο και περισσότερε ανθρώπινε ζωέ. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε πολύ πιο αποτελεσματικά και να μειώνουμε επίσης και τις δαπάνες επέμβασης διάσωσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιστοποιήσουμε την οδική ασφάλεια. Και υπάρχει και άλλη μια άλλη πτυχή πολύ σημαντική, το ζήτημα της ευελιξίας, Το ότι προβλέπονται δηλαδή οι δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών υποδομών οι οποίες όπως και το σύστημα e θα σέβονται την ιδιωτική ζωή και τα, ανθρω... και τα προσωπικά δεδομένα. Όπως ακούσατε όλα αυτά τα δεδομένα θα διαγράφονται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες αναφέρονται περισσότερο στα προσωπικά δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα θετικότατο μήνυμα προκειμένου να καταφέρουμε να εγκρίνουμε το νέο αυτό σύστημα το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Για 1,5 λεπτό, εκπρόσωπος των φιλελευθέρων, η κυρία Κάλασα. Η ψηφοφορία αυτή είναι το τελευταίο βήμα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα αυτό θα εγκαθίσταται σε όλα τα οχήματα στην Ευρώπη. Ε, χαίρομαι που περιλαμβάνονται καινούς διατάξεις που διασφαλίζουν ότι δεν θα τύχαν κατάχρησης και ότι θα προστατεύεται η ιδιωτική ζωή. Η ιδιωτική ζωή των ατόμων είναι πολύ σημαντική. Ο στόχος του ΕΚΟΛ είναι να σώζει ζωές και θα πρέπει να περιοριστεί σε αυτή τη λειτουργία. Να θυμηθούμε ότι οι ζώνες ασφαλείας μείωσαν τον αριθμό των ε, θυμάτων κατά 40 περίπου της 100 παρόλο ότι όταν αποφασίστηκε η χρήση τους ε, πολλοί ήταν διστακτικοί. Μετά είχαμε το airbag, τον αερόσακο και τώρα έχουμε το e-call. Προφανώς ε, χρειάζεται να αλλάξουμε συνήθειες, να εμπιστευτούμε τη νέα τεχνολογία αλλά τεχνολογίες όπως το e-call μπορούν να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Σε χώρες όπως η Εστονία με πολλή ε, κυκλοφορία στους δρόμους ε, θα είναι χρήσιμο ε, να καλούνται αμέσως οι υπηρεσίε διάσωσης. Να πω επίσης στους συναδέλφους που είπαν ότι το σύστημα είναι ελεύθερο, πως ένα σύστημα ποτέ δεν είναι ελεύθερο, ε, δωρεάν, συγγνώμη, δεν είναι δωρεάν, διότι υπάρχει ένα κόστος επένδυσης, οπότε αυτό θα αντικατοπτριστεί στις τιμές. Παρ' όλα αυτά θα εξασφαλίζει αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εξ ονόματος της ε, Γκουε, η κυρία Κιούλενεν. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Μικρόφωνο σας. Συνάδελφοι, το σύστημα e-call θα αποτελέσει προηγούμενο, ε, διότι στο μέλλον θα πρέπει να δώσουμε όλο και περισσότερο βάρος στην, ε, στη ρύθμιση του, της οδικής κυκλοφορίας, ε, στην συλλογή και μετάδοση πληροφοριών κλπ. Δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε κατά περίπτωση να νομοθετούμε για αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να ορίσουμε κάποιες αρχές, κάποιες κόκκινες γραμμές ε, και μετά να κινηθούμε ανάλογα ομάδες είναι διχασμένες εδώ στο Κοινοβούλιο. Να θυμηθούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είμαστε ταγμένοι στην ε, μείωση ε, των θυμάτων από τα ατυχήματα κατά 50%. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Ο αριθμός των θυμάτων αυτή τη στιγμή είναι περίπου 27.500 το χρόνο. Μια μικρή πόλη δηλαδή ενδιαφέρομαι για αυτά τα θέματα και δεν μπορώ να δεχτώ ότι η προστασία των ατόμων και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ανταγωνιστικά πράγματα. Όχι, θα πρέπει να τα φροντίσουμε και τα δύο. Θα πρέπει αυτό να συμπεριληφθεί στην ψηφιακή ε, ατζέντα κυκλοφορίας. Ευχαριστούμε εξ των Πρασίνων για 1,5 λεπτό κύριο Σάλμπρεχτ. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Σάλμπρεχτ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και για το πολύ καλό έργο της σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Κατανοώ ότι υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση των πληροφοριών που διαβιβάζονται από το σύστημα, αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Το σύστημα e-call δεν πρόκειται να αποτρέψει κανένα ατύχημα. Οι ασφάλεια στους δρόμους και η πρόληψη των ατύχημάτων έχουν να κάνουν με το να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του προβλήματος αυτού, όπως χάρη υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσει να μειωθεί πραγματικά ο αριθμός των ατυχημάτων. Προφανώς το e-call θα βοηθήσει σε ταχύτερη έλευση των σωστικών ε, συνεργείων αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί το θέμα του κάτω από ποιες συνθήκες, με ποια ιδιότητα θα στείλει αυτό το σύστημα. Το να έχει κανείς το σύστημα e-call ως οδηγός ενός αυτοκινήτου είναι θετικό. Γιατί όμως να μην έχει τη δυνατότητα αυτός ο οποίος αγοράζει ένα αυτοκίνητο να δίνει και τη συγκατάθεσή του για αυτό το σύστημα να λέει ναι το θέλω ή δεν το θέλω αυτό το σύστημα. Γιατί αυτό το οποίο βρίσκεται μέσα σε αυτό το κουτί είναι μια σύνδεση κινητής ε, τηλεφωνίας και εάν θέλει το σύστημα να πάρει πληροφορίες για το πού βρίσκεται ένα όχημα, μπορεί μέσω του συστήματος αυτού να αποκομίσει τις πληροφορίες. Δεν θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί της πανδώρας και να επιτρέπεται να υπάρχει παρακολούθηση και ανήφθεση σε αυτοκίνητο που και να είναι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάιερ, μη εγγεγραμμένος, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και για μένα αυτή η εφαρμογή του συστήματος e-call είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε θετικά. Δεν είναι κάτι το απόλυτα καινούριο. Υπάρχει ήδη σε διάφορους ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων ένα αντίστοιχο σύστημα. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να αποτρέψει τα ατυχήματα όπως ελέγχει αλλά μπορεί να κερδίσει πολύτιμο χρόνο μεταξύ του ατυχήματος και της παρουσίας των σωστικών δυνάμεων. Παρά όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν μερικά προβλήματα που δεν έχουν επιληθεί. Ένα από αυτά είναι ότι οι κατασκευαστές οι οποίοι έχουν ήδη ένα σύστημα θα πρέπει να εγκαταστήσουν και το δεύτερο αυτό σύστημα. Επίσης νομίζω ότι είναι κάπως αισιόδοξη η προθεσμία που αναφέρεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2017. Πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ακριβώς όπως αναφέρθηκε η προστασία των δεδομένων και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις που έλαβαν χώρα και πολλές ανάγκες να υπάρξει περαιτέρω διαλεύκανση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 μπορεί κανείς να συζητήσει για πολλά θέματα, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή παίρνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων των οδηγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χαίρομαι για το γεγονός αυτό και χαίρεται ιδιαίτερα και η ομάδα του ΕΛΚ. Αύριο στη δεύτερη ανάγνωση υπάρχει μοναχα μία τροπολογία και αν θυμάμαι καλά είναι από τους φιλελεύθερους. Οι φιλελεύθεροι όμως δεν έχουν ε, επιχειρηματολογήσει για αυτό το θέμα και τίθεται και το θέμα και από τους πράσινους είναι το ζήτημα της προστασίας δεδομένων. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να στέλνετε η κλήση στο 112 μόνο όταν ενεργοποιηθεί ο αερόσακος. Μπορεί να γίνεται αυτό όταν υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα μέσα στο αυτοκίνητο και όχι μονάχα με τον αερόσακο. Νομίζω ότι η συμβαστική λύση που ευρέθη σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και η ανάγκη για τη βελτίωση της ε, υποδομής για την, ε, ε, τη διάσωση έκτακτης ανάγκης είναι πάρα πολύ σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μονάχα το θέμα λοιπόν της οδικής ασφάλειας, αλλά το να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει υποδομή σε όλα τα κρατημέλη, ώστε οι κλήσεις του 112 να καταλήγουν. Κύριε Σφάμπα, υπάρχει μία μπλε κάρτα για σας, την αποδέχεστε. Εξ ονόματος του κύριου Ρούμπικ. Κύριε Ρούμπικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζλούμπη. Αγαπητέ συνάδελφε Σουάπ, θα ήθελα να ξέρω... Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι από τεχνική έποψη είναι έτοιμο και όριμο το σύστημα αυτό το εικόν για να εφαρμοστεί στα οχήματα. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Είμαστε στη δεύτερη ανάγνωση και είναι απαραίτητο όχι μόνο να λειτουργεί πλήρω το σύστημα 112, αλλά και να παραμείνουν και τα ιδιωτικά συστήματα οδική βοήθειας. Τίποτα όμως δεν πρέπει να εμποδίσει να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο 112 και να υπάρξει η τυποποίηση για τον τρόπο πρόσβασης. Αυτό θα ωφελήσει όλους. Ο Χόλσερ, λεπτό παρακαλώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια, την κυρία Σέχνάλοβα, για την πολύ καλή εργασία της. Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι με, αυτή την, ε, με αυτόν τον κανονισμό μπορούμε να διασώσουμε περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Για μένα είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει βρει μια κοινή θέση η οποία βελτιώνει την αρχική πρόταση της Κομισιόν και αυτό καταδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο και οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ του. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο επίση πρέπει να λεχθεί και να το χαιρετήσουμε. Τέλο, θέλω να σταθώ και εγώ στο θέμα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Έχουμε ήδη συζητήσει πάρα πολλά για την συγκατάθεση ή όχι σε σχέση με την απόστολη των δεδομένων αυτών. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε μια καλή λύση η οποία εξασφαλίζει τις βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων και εν κατακλείδη θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι προσβάσιμο από όλους και έχει οικουμενικό χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο έχει ο Ντάλτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόληψη των ε, τροχαίων ατυχημάτων είναι πολύ σημαντική και την υποστηρίζουμε, όμως θα πρέπει να εστιάσουμε στις στρατηγικές και τους μηχανισμούς που είναι πιο αποτελεσματικοί για την, αύξηση της ασφάλειας. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να δεχτώ την υποχρεωτική εγκαταστήση αυτού του συστήματος για τέσσερις λόγους. Πρώτον, διότι χρησιμοποιούνται, ε, χρησιμοποιούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που δεν υπάρχουν παντού. Ιδιαίτερα στο ΕΒ. Βασίλειο. Ε, δεν θα λειτουργεί εκεί που το σήμα δεν είναι ισχυρό. Δεύτερον, χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές ε, παρόλο ότι η μείωση θα είναι 0,5% στα θανατηφόρα ατυχήματα. Χρειάζεται καλύτερα λοιπόν να βελτιώσουμε τις υποδομές, τις οδικές υποδομές. Ε, τρίτον, έχουμε ενισχύσει ό,τι αφορά την ιδιωτική ζωή. Ε, δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις των οχημάτων μέσα αυτού του συστήματος. Είναι απαράδεκτο το σύστημα θα πρέπει να είναι θελοντικής χρήσης και εγκατάστασης, όχι υποχρεωτικής. Μόνο ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Μάισνερ για ένα, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Σεχνάλοβα για την εργασία της και τη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους. Σε ένα σημείο μπορώ να συνδεθώ με αυτά τα οποία είπε ο προλαλής Είναι πολύ καλό το σύστημα η e γιατί μπορεί να βοηθήσει τις σωστικές διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήματος. Αλλά το θέμα για μένα είναι το εξής, να πάρει το να έχουμε καινοτομίε στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Αλλά όλα αυτά εμπλέκονται στα θέματα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ξέρει κανείς ο οδηγός αν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει μόνο το σύστημα και αν πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες για να αποφύγει την ε, παράδοση προσωπικών δεδομένων. Αλλά αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν από μόνα τους. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν αν Θέλει κανείς να χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα ή όχι. Είναι ένα θέμα για την προσωπική σφαίρα των Ευρωπαίων πολίτων. Γι' αυτό εγώ θέλω να υποστηριχθεί η τροπολογία των φιλελευθέρων που κινείται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ πολύ γιατί ήταν πολύ σύντομοι και κερδίσαμε χρόνο. Η κυρία Τροζίνσκη τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η οδική ασφάλεια χάρη στη σύσταση αυτή ε, είναι, γίνεται θέμα προτεραιότητας. Στην ε, Γαλλία η ε, οδηγία είναι πολύ ευαίσθητη για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, πολλοί λένε ότι θα είναι δωρεάν η χρήση του πλην όμως θα υφίσταται ένα κόστος για την άνθρωση της υποδομής κάτι που θα αντικατοπτριστεί στην τιμή του, του οχήματος. Ε, τι κάνει αυτό το σύστημα, καλεί το 112 και στέλνει και ένα σήμα GPS. Ε, οι πρόθεσει είναι καλές, αλλά η ανάλυση αντικτύπου που υποβλήθηκε είναι, δεν είναι πιστική. Ε, ελάχιστη η μείωση των θανάτων, 10 ε, 15% η μείωση των τραυματισμών. Έχουμε μιλήσει επί μακρόν για θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικής ζωής. Αυτό είναι που μας ενισχύει περισσότερο. Πώς θα μας εγγυηθείτε ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα ε, τύχουν εκμετάλλευσης για διαφορετικούς λόγους. Ε, το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε, να προστατεύσουμε την ε, οικονομική κατάσταση των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γκαλπέλτς για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, καταρχήν να πω ότι η δυνατότητα ε, ε, να παράσχεται άμεση βοήθεια σε τέτοια ατυχήματα είναι αναπόσπαστο βήμα της εσωτερικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί η δουλειά της ήταν πραγματικά εξαιρετική. Σας υπενθυμίζω ότι καταρχήν είχε δημοσιευθεί ένα ψήσιμο το 2012 από τότε δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ήταν οι με εμπειρογνώμονες, οι παρουσιάσει κλπ. Αμέτρητε. Όλοι προσπάθησαν πολύ. Σε μια κατάσταση εκτέκτης ανάγκης είναι σημαντικό να διαθέτουμε ένα σύστημα υποχρεωτικό που να μην μπορεί μάλιστα κανείς να το σβήσει από μόνος του. Να το θέσει εκτός λειτουργίας. Για παράδειγμα, ένας οδηγός μπορεί να έχει τραυματιστεί, να έχει χάσει τις αισθήσει του. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα. Είναι σημαντικό το σύστημα να είναι ενιαίο για όλους, υποχρεωτικό σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία του, δωρεάν στη χρήση του και ε, να υφίσταται σε όλα τα κράτη-μέλη. Κατανοώ ότι η επένδυση δεν είναι φτηνή, γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό οι επενδύσεις να γίνουν με ομοιογενή τρόπο και το σύστημα αυτό να είναι παρόν σε όλα τα οχήματα. Μέχρι το 2018 έχουμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να ρυθμίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου το σύστημα να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία. Το σύστημα αυτό πιστεύω θα σώσει τη ζωή δεκάδων χιλιάδων ατόμων. Το δικό μας καθήκον είναι να το αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Στήλερ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Όλκα Σενάλοβα για την εξαιρετική της εργασία ήδη από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία μέχρι σήμερα. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά καταβλήθηκαν σημαντικότερε προσπάθειες και έχουμε μια εξαιρετική πλέον πρόταση νομοθεσία που θα σώζει χιλιάδες ζωές στη Σκωτία, τον Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Η οδική ασφάλεια μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση ατυχήματος θα ενεργοποιείται αυτόματα ένα σύστημα το οποίο θα ειδοποιεί τι ομάδε διάσωση και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πολύ καλύτερα όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε και οι οικογένειε οι οποίε ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω του συστήματο αυτού να αυξήσουμε την ποιότητα τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και το βλέπουμε πλέον αυτό με όλε αυτέ τι ευφυεί υπηρεσίε, με το λεγόμενο ίντερνετ των πραγμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο η ηλεκτρονική ασφάλεια, το e-safety αλλά και το σύστημα e-call αποτελούν τον, τη νέα αυτή δέσμη, νέε τεχνολογίε που θα πρέπει να έχουμε καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα αυτά αντικείμενα, τα νέα προϊόντα και τι νέε εφαρμογέ, τι οποίε τι βλέπουμε πλέον να αντικατοπτρίζονται στη νέα αυτή πρόταση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Φόρντ για ένα λεπτό. Nearly people die in... 26.000 άτομα πεθαίνουν σε οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Αν έχετε βρεθεί με το αυτοκίνητό σας αναποδογισμένο με όλη την οικογένειά σας, όπως βρέθηκα εγώ πέρσι το καλοκαίρι, και θέλετε να σας φτάσουν τα σωστικά συνεργεία το ταχύτερο δυνατό, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπήρξαν φυσικά ανησυχίε για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα και αντιμετωπιστήκαν ορισμένα θέματα στις ε, συζητήσεις του τριγωνικού διαλόγου. Και βέβαια είναι κάπως παρεμβατικό το να έχετε κάτι μέσα στο αυτοκίνητό σας το οποίο δεν μπορείτε να το σβήσετε όπως ένα μικρόφωνο. Ίσως θα έπρεπε να είναι πιο εθελοντικού χαρακτήρα αυτό το μηχάνημα και είναι κάπως αποκλειστική η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται και εγώ ανησυχώ που δεν αφήσαμε τη δυνατότητα να υπάρξουν άλλες ευφυείς και ενωτόμες πρωτοβουλίες. Θα είναι ακριβό το σύστημα αυτό, 100 ευρώ και παραπάνω ανά αυτοκίνητο, αλλά κυρίως θα είναι υψηλό το κόστος της υποδομής που θα το υποστηρίζει. Δυστυχώ τα χρήματα αυτά ε, αποσπούνται από άλλα μέτρα διάσωση Μου λένε οι εμπειρογνώμε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο για τη βελτίωση των οδικών συστημάτων ή για περαιτέρω έρευνα, ότι, ώστε τα αυτοκίνητα να μην αναποδογυρίζουν. Για αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι η συγκίτρια έχει κάνει πολύ καλή εργασία για να βελτιωθεί αυτό το νομοθέτημα, πιστεύω ακόμα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ευφυή, ε, καλύτερη και πιο εθελοντική λύση. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Πρέπει να σας πω ότι καθότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη από τις εννιά εκθέσεις που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα, δεν είναι δυνατόν να πάρετε όλοι το λόγο όσοι συζητήσατε να πάρετε το λόγο στα πλαίσια του Catch the Eye. Οκτώ μόνο άτομα, οκτώ ευρωβουλευτές μπορούν να πάρουν το λόγο, εκπροσωπώντας βέβαια τις πολιτικές τους ομάδες. Η κυρία Τούν Όινστάιν έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ στηρίζω την υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση του ε, συστήματος αυτού σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα. Ε, σε όσους το φοβούνται να υπενθυμίσουμε και να επαναλάβουμε ότι καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα κατάλληλο και παρκές επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής ε, Κανείς δεν θα μπορεί να παρακολουθεί, να εντοπίζει την πορεία ενός οχήματος με αυτό το σύστημα ε, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό Πρόκειται για θέματα ασφάλειας, πρόκειται για θέματα ανθρώπινης ζωής. Και σίγουρα έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Απομένουν πολλά ακόμα για να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Χρειάζεται, για παράδειγμα, να μειώσουμε ακόμα και την μόλυνση που προέρχεται από τα ε, να, να βελτιώσουμε και τα συστήματα ε, φίλτρων ε, που περιλαμβάνονται στα συστήματα μείωση των εκπομπών. Ε, οπότε έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να προσέξουμε στο μέλλον. Η ασφάλεια, η οδική ασφάλεια θα εξαρτηθεί από το πόσο προσεκτικοί θα είμαστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι ο χρόνος ο οποίος χρησιμοποιείται για την οδική διάσωση έχει να κάνει βέβαια με την ίδια τη διατήρηση των ανθρώπων στη ζωή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία αυτή που έχουμε πλέον για το e-call, για τα νέα οχήματα και για τα ελαφριά οχήματα αποτελεί ένα σημαντικότατο ε, βήμα πρόοδου για την προστασία της ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Να ευχαριστήσω την κυρία Σενάλοβα και τους εκπροσώπους Ιταλικής Προεδρίας, ε, διότι προώθησαν το ζήτημα αυτό με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα, προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό κανονισμό σε συγκεκριμένα πρότυπα οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι εμπλέκονται στο σύστημα αυτό πάρα πολύ διαφορετικοί κλάδοι και εμπλέκονται και πολλέ διαφορετικέ πτυχέ που έχουν να κάνουν από τη μια με την οδική ασφάλεια και από την άλλη με την προστασία τη ιδιωτικής ζωή. Απαιτούνται συνεχώ όλο και υψηλότερα πρότυπα και προδιαγραφέ. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών θεωρώ ότι έχουμε βρει μια καταπληκτική συμβαστική λύση. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα πραγματικό παράδειγμα το ότι η ολοκληρωμένη Ευρώπη μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένε αποφάσει για την προστασία των πολιτών τη. Τέτοιε αποφάσει χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο και ελπίζω πραγματικά ορισμένοι συνάδελφοι που το είπαν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να μην καταφέρουν να αποδυναμώσουν μια πρόταση που τελικά αυξάνει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Κόρμπετ διαδικαστικό, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ούτε ένας ομιλητής από την ομάδα του EFTD ε, ε, γιατί πιστεύει το EFTD ότι δεν είναι καλή νομοθεσία ή γιατί βρίσκονται σε αμηχανία που βλέπουν ένα νομοθετικό κείμενο που στηρίζεται τόσο πλατιά. Ε, Κοιτάξτε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η πολιτική ομάδα του EFDD δεν ζήτησε να πάρει το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Περνάμε στη δικασία Catch the Eye. Η κυρία Παουνόβα για ένα λεπτό παρακαλώ. Η αυριανή ψηφοφορία για την ανάπτυξη του συστήματος e-call, λέει η κυρία Πάουνοβα, δεν είναι μονάχα το επιστέγασμα έξι και πλέον ετών προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκπροσωπεί επίσης και μια παρότρεση προς τη Κομισιόν να υποβάλει νομοθετικά μέτρα του ταχύτερο δυνατό, ώστε το σύστημα e-call να είναι υποχρεωτικό σε όλες τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. μέχρι το 2018. Η αυριανή ψηφοφορία όμως είναι και ένα αποφασιστικό βήμα για να εδραιώσουμε την ύπαρξη ενός συστήματος το οποίο μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πώς και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσθέσει αξία για τους πολίτες της. Με αυτές τις ε, εξελίξεις που, όπου παίζει σημαντικό ρόλο και η ψηφιακή τεχνολογία η διασυνδετικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά πολλά θέματα, αλλά μας ενδιαφέρει πάντα και η προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Υπήρξε λοιπόν σημαντική μνήμα για τις προσωπικές, τα προσωπικά στοιχεία, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματο και όχι για την παρακολούθηση των οχημάτων. Κάνω μια έκκληση πώ λοιπόν, θα κάνει μέλη και στου αυτοκινητοβιομηχάνου να κάνουν το απαραίτητο να εφαρμοστεί το σύστημα ταχύτερα δυνατό. Κυρία Φλασικόφα Μπενόβα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ζήτημα αυτό είναι προφανώς ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ωστόσο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Όλκα Σενάλβα, γιατί κατάφερε πραγματικά να συντάξει μια εξαιρετική έκθεση. Ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό από το 2005. Θεωρώ λοιπόν ότι το καινοτόμο αυτό σύστημα κλήσης έκτατης ανάγκης, ε, e-call, θα σώσει χιλιάδες ζωές και είναι πραγματικά κρίμα το ότι μετατέθηκε η ημερομηνία θέση σε ισχύω του κανονισμού αυτού. Η ε, οδική ασφάλεια θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο καθυστερούμε την εφαρμογή ενός κανονισμού που θα σώσει όλο και περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Τα στατιστικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα θλιβερά. Μολονό, αυξάνοντα λοιπόν την, οδική ασφάλεια, την ενεργή οδική ασφάλεια, θα πρέπει να αυξήσουμε παράλληλα και την παθητική οδική ασφάλεια και θα πρέπει να αυξήσουμε και την αποτελεσματικότητα των διασωστικών ομάδων και συνεργείων. Θεωρώ λοιπόν ότι το νέο αυτό σύστημα e-call θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα και ότι θα βοηθήσει στο να διασωθούν ζωές στα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Ξέρετε ότι κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό μετράει και είμαι πεπισμένος ότι, πληροφορίες, ότι το ζήτημα αυτό τελικά θα βοηθήσει πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες. Να αμφισβητήσει τη χρησιμότητα του συστήματος του e που πραγματικά θα μπορέσει να σώσει ζωές μετά από τροχαία ατυχήματα. Να συμβάλλει έτσι στην ασφάλεια ε, κατά τη διάρκεια των ε, μεταφορών. Όμως το θέμα είναι ποιες οι εγγυήσει για τα προσωπικά δεδομένα. Ποιες οι εγγυήσει για να μην υπάρχει έλεγχος της ιδιωτικής ζωής νομίζω ότι από τη συζήτηση προέκυψε ότι δεν υπάρχουν πλήρεις εγγυήσεις. η περίφημη αρχή της ευελιξίας δημιουργεί ένα σημαντικό κενό. η διατήρηση δεδομένων έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα νομίζω ότι αποτελεί μια απαρχή όπου ενδεχόμενα με μια τροποποίηση του κανονισμού στο μέλλον να διατηρούνται τα στοιχεία αυτά και για πολύ περισσότερο διάστημα δεν μας εξηγήθηκε τι σχέση έχει αυτή η σημαντική πράγματι υπηρεσία με την λεγόμενη ψηφιακή κυκλοφορία και τις επιλογές οι οποίες θα γίνονται. δεν μας ενημέρωσε κανείς για το πώς αυτό το σύστημα θα λειτουργεί με την περίφημη αυτόματη κυκλοφορία των οχημάτων στο μέλλον. όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν για να υπάρχουν οι εγγυήσει στην ιδιωτική ζωή και για να μην γίνεται παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκοβιτς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ελέγχθη ότι το σύστημα αυτό είναι οικονομικό, ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο. Σύστημα το οποίο μπορεί να σώσει ζωές. Τις ζωές των οδηγών και των επιβατών οχημάτων. Υπερβολικά πολλοί συμπολίτε μα χάνουν τη ζωή τους ε, στην άσφαλτο. Το γεγονό ότι βοήθεια θα φτάνει πιο σύντομα θα μειώσει τον αριθμό των θυμάτων όπως έγινε και με τις ε, ζώνες ασφαλείας, όπως έγινε και με τους αερόσακους. Ως ε, μέλος της ομάδας μου Μπορώ να σας πω ότι ήταν σημαντικό για την ομάδα μας ε, να υπέλθει συμφωνία για το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Και αυτό υποστηρίζω ε, και ψηφίζω θετικά για την εγκατάσταση του συστήματος. Σέλτες. Σέλτες, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ασφάλεια στις, ε, στους δρόμους μας είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων στους δρόμους κάθε χρόνο. Αναφέρθηκε ο αριθμός των 26.000 νεκρών το χρόνο. Και συγχρόνως είναι απαραίτητο να κάνουμε περισσότερα και για την πρόληψη των ατυχημάτων στους δρόμους, ώστε να υπάρξει μια μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας κατά 10 χιλιόμετρα που μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση των θανάτων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει όχι μοναχά μια εξτατεία για την πρόληψη αλλά και για την καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών. Επίσης να ε, εμποδιστεί η οδήγηση οδηγών που έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Το μέτρο του e-call δεν πρόκειται να σταματήσει βέβαια τα ατυχήματα στους δρόμους, αλλά θα μειώσει τον αριθμό των θαμάτων. Είναι απαραίτητο να γίνουν σωστές λύσεις όμως και για την προστασία των δεδομένων. Κύριο Σόμπερ Μάια κύριε Πρόεδρε. Ένα αυτόματο σύστημα έκτακτης κλίσης με ταχεία ε, προσέλευση των σωστικών συναρχείων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι πολύ θετικό, αν είναι διαθέσιμα τα σωστικά συνεργεία. Υπάρχει όμως και η ανάγκη να υπάρξει προστασία των δεδομένων των οδηγών. Αν υπάρχει μία πληθώρα στοιχείων όπως θα ζητήσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αυτό δεν πρόκειται να είναι καλό. Δεν πρέπει επίσης να δώσουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια απατηλή έννοια, ε, αντι, μάλλον εντύπωση ε, προστασίας. Γιατί όλα εξαρτώνται από το πόσο διαθέσιμες είναι οι δυνάμεις διάσωσης. Δεν πρέπει λοιπόν να παραπλανηθούν οι οδηγοί για το πόσο γρήγορα μπορούν να διασωθούν. Υπάρχει πολύ έργο ακόμα το οποίο πρέπει να γίνει για να μπορέσει να εξασφαλιστεί αυτή η έγκαιρη διάσωση σε όλη την Ευρώπη, ιδίως σε χώρες όπως η Αυστρία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαριάννα Πέτυρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το Κοινοβούλιο στήριξε την εισαγωγή του συστήματος e ε, με τον κανονισμό αυτό ε, το σύστημα αυτό θα εγκατασταθεί σε όλα τα ε, οχήματα και θα σώνει ζωές ε, προστατεύοντας ταυτόχρονα τις προσωπικές πληροφορίες. Το σύστημα αυτό καλεί αυτόματα τον αριθμό 112 σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιείται δωρεάν. Βέβαια, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ε, θα, και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διοργανώσουν εκστρατείες ε, για την ενημέρωση των καταναλωτών για το πόσο σημαντικό είναι το σύστημα αυτό. Ε, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολιτές να μπορούν να εντοπιστούν σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ε, θα πρέπει να ε, ε, βελτιώσουμε και τις υποδομές για να συμβεί στο μέλλον. Πάντως είναι σημαντικό να εγκατασταθεί το σύστημα αυτό, το οποίο θα λειτουργεί αυτόματα και θα καλεί το 112. Καπούτο, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το σύστημα αποτελεί σημαντική βελτίωση και συνδέεται επίση και με τα άλλα συστήματα, τα ιδιωτικά και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια. Μπορούμε μέσω του συστήματο αυτό να βοηθήσουμε πάρα πολύ γρήγορα του οδηγού οι οποίοι εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σώσουμε εκατοντάδε και χιλιάδε ζωέ κάθε χρόνο. Μέσω τη αποστολή συγκεκριμένων δεδομένων όσον αφορά το γεωγραφικό εντοπισμό ενό οχήματο, μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να διασώσουμε όλο και περισσότερου ανθρώπου πολύ πιο αποτελεσματικά και γρήγορα. Ωστόσο, σημαντική προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί και στην ιδιωτική ζωή καθώς επίσης και στην συλλογή και την διατήρηση των δεδομένων αυτών σε δημόσιες αρχές και όχι σε, ιδιωτικές, σε ιδιωτικούς φορείς. Τα δεδομένα αυτά, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανταυτού προκειμένου να καταφέρουμε να χειριστούμε καλύτερα την κίνηση στους δρόμους των, ευρωπαϊκών πόλεων. Ο κύριος Χόγκαν έχει το λόγο. Κύριε Χόγκαν, έχετε το λόγο και ολοκληρώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στη συζήτηση για το επικοδομητικό πνεύμα διαλόγου ήταν πολύ θετικό να έχω την ευκαιρία να ακούσω όλα αυτά τα μέλη τα οποία θα αναλάβουν το λόγο για το ζήτημα αυτό. Η συζήτηση έκανε σαφές ότι υπάρχει συντριπτική υποστήριξη για το σύστημα e-call και χαίρομαι για αυτήν την υποστήριξη. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταδείξει την αποφασιστικότητά του και την υποστήριξη για το να υλοποιηθούν τα ωφέλη του συστήματος e-call. Και είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει μια μεγάλη, ένα μεγάλο επίπεδο συνένεσης για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Δεν είναι ένα θέμα μονάχα ε, τεχνολογίας ε, που εγκαθίσταται στα αυτοκίνητα. Είναι κυρίως θέμα τεχνολογίας για να προσδιορίζεται και να αναφέρεται η ακριβής θέση ενό οχήματο που έχει υποστεί ατύχημα. Δεν είναι θέμα λοιπόν για προσωπικά δεδομένα. Εστιάζει στο να σωθούν οι ζωέ οι οποίε εμπλέκονται σε ένα ατύχημα. Φυσικά τα ατυχήματα θα συμβαίνουν δυστυχώ πάντα λόγω της συμπεριφορά των οδηγών. Αλλά δεν πρόκειται να αποστερηθούν πόροι από τις προσπάθειες αύξησης της οδικής ασφάλειας μόνο και μόνο γιατί η τεχνολογία για το σύστημα γίνεται πια ένα τμήμα της ε, διαδικασίας ε, παραγωγής αυτοκινήτων. <clears throat> Ξέρω ότι η κυρία Βίκη Φόρτ είχε ανησυχίες σε σχέση με το κόστος προς τον καταναλωτή με την εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι τα 100 ευρώ είναι <clears throat> οι πιο υψηλές εκτιμήσεις σε σχέση με το κόστος αυτών των συστημάτων γιατί τα συστήματα χρήσης κινητών τηλεφώνων και GPS υπάρχουν ήδη σε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Επομένως είναι πολύ μικρό το κόστος για να προσθεθεί και αυτή η τεχνολογία στο στάδιο της κατασκευής των αυτοκινήτων ώστε να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια, τους και εισηγητές και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολύ θετική συζήτηση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει η εισηγήτρια η κυρία Σενάλοβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν στη συζήτηση αυτή, και οι οποίοι είπαν ότι υποστηρίζουν την πρόταση αυτή και υποστήριξαν την πρόταση αυτή σε όλη την νομοθετική της πορεία. Όπως το είπα ήδη, Είχα ακούσει κάποιε επικριτικέ παρατηρήσει στην αρχή όσον αφορά το σύστημα αυτό. Τώρα όμω είμαι πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια των κρατών μελών κατάφερε τελικά να λάβει υπόψη του στο κείμενο αυτό όλε αυτέ τι παρατηρήσει και τις επικρίσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πεπισμένη ότι η ανάπτυξη του συστηματο e e-call στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στη βελτίωση τη ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου παντού στην Ευρώπη. η μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και των θανάτων στο δρόμο αποτελεί πραγματική προσδοκία, πραγματική επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αυριανή λοιπόν ψηφοφορία θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τον στόχο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται η ζήτηση από το σημείο. Η ψηφοφορία θα δεξαχθεί αύριο.